να συνεχίζουμε ανεξαρτήτως των συνθήκων που επικρατούν, όσο δύσκολες και αν είναι αυτές. Ναι, ναι, δεν πρέπει να αποθαρρυνόμεθα, πράγματι λέει ο Πρόεδρος.